ασθενεί ή οροθετικοί ασθενεί του. Και η κοινωνία θα ε, πρέπει να μπορεί να προστατεύεται, όχι μόνο οι άρρωστοι. Ευχαριστώ.